Okay, I think um, we can now. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την ακρόαση για τον διορισμό του Προέδρου της, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας. Υπάρχει μερίσια διάταξη με ένα βασικό σημείο, δηλαδή η ακρόαση, δεν νομίζω να έχει κανείς σας αντίρρηση. η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε θα είναι η σύνηθις διαδικασία, δηλαδή η Ντανιέλ Νουή θα κάνει μία σύντομη παρουσίαση 10 λεπτών και μετά <clears throat> έχουμε ήδη έναν κατάλογο ομιλητών που θα θέσουν κάποιες ε, ερωτήσεις. Πέντε λεπτά ο καθένας. Προσπαθήστε να είστε λογικοί, να μην κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί προφανώς ε, δεν ε, θα μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, εάν είναι πολλές, πρόκειται για μια ακρόαση, έτσι, να είστε λογικοί. Ντανιέλ, θα ήθελα να σε καλωσορίσω και να σου δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που απευθύνομαι σε αυτή την ακρόαση εδώ σε εσά μετά από την ε, υποψηφιότητά μου που έγινε δεκτή σαν υποψήφια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα να ε, παρουσιάσω και να υπογραμμίσω την εμπειρία που έχω ε, στα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των τραπεζικού συστήματος. Όλη μου η καριέρα έχει αφιερωθεί στα θέματα της ε, τραπεζικής εποπτείας και τραπεζικού ελέγχου και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο και σε περιόδους ηρεμίας και σε περιόδους κρίσης. Τα τελευταία δέκα χρόνια είμαι υπεύθυνη της ε, επικεφαλής της του γαλλικού εποπτικού τραπεζικού συστήματος. Την ίδια περίοδο, τα τελευταία δηλαδή δέκα χρόνια, έχω αναμειχθεί ενεργά στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 με την ε, ε, Επιτροπή Επαφής και μετά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, της για την τραπεζική εποπτεία. Είμαι μέλος του Συμβουλίου και της ΕΜΠΑ και της ΕΙΟΠΑ. Έχω εκλεγεί και στο Διευθυντικό Συμβούλιο των δύο αυτών αρχών. Ας ε, δούμε τώρα ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει το τραπεζικό μας ε, σύστημα και το κυρίως το τραπεζικό, το ενιαίος μηχανισμός μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης της κρίσης πιστεύουμε ότι η τραπεζική εποπτεία θα βοηθήσει τον Ευρωπαίο πολίτη ε, και πιστεύουμε ότι η Τραπεζική Ένωση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών μας. Το, ο ενιαίος αυτός ο μηχανισμός, ο εποπτικός μηχανισμός στηρίζεται στα όσα έχουν γίνει ε, στα θέματα τραπεζικής εποπτείας Έχουμε διάφορα σημαντικά στοιχεία και διάφορες αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν και που, όπου ε, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ήταν ζωτική σημασίας. Και έχει δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή κουλτούρα εποπτείας με όλη αυτή τη διαδικασία. ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας θα συνδυάζεται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εποπτείας, με την ΕΜΠΑ πιο συγκεκριμένα και είμαι σίγουρη ότι ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας θα είναι προς όφελος της ΕΜΠΑ και θα αλληλοστηρίζονται κυρίως όσον αφορά τον, τους ενιαίους κανόνες ε, ο ορισμός όσον αφορά την, τα, τα δάνεια και τα, τα, τα, τα stress test των, τραπεζών. Τώρα, για το, το ενιαίο σύστημα, ο μηχανισμός εποπτείας, πιστεύουμε ότι θα γυρίσει μια νέα σελίδα στην Ευρώπη, θα σέβεται τον διαχωρισμό ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και στην τραπεζική εποπτεία. Ο ενιαίος μηχανισμός θα στελεχωθεί από ελεγκτές, από επόπτες ε, που θα έχουν τα ε, ύψιστα προσόντα αν θέλετε και θα εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει να ε, ακολουθήσει και να εφαρμόσει την, την εποπτεία με, τους καλύτερα, με τα καλύτερα δυνατά στελέχη και πραγματικά θα πρέπει να τονίσουμε την ποιότητα τις εποπτείες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις καλύτερες εποπτικές πρακτικές οπουδήποτε και βρίσκονται αυτές και να τις εφαρμόσουμε. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε και καινοτόμοι, να βρούμε και καινούριε ιδέες. Η ποιότητα της εποπτείας και του ελέγχου ε, εξαρτάται επίσης και από το γεγονός ότι η ΕΚΤ θα είναι η μοναδική επόπτης, αν θέλετε, όλων των τραπεζών σε όλη την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Άρα θα υπάρχει μια σύγκληση των πολιτικών εποπτείας. Και ε, το, το γεγονός ότι θα υπάρχει η ΕΚΤ ε, προφανώς θα αποτρέψει από τον πειρασμό ε, να εφαρμοστούν εθνικές πολιτικές. Επίσης, θα, οι επόπτες θα είναι ανεξάρτητες, σε σχέση με, την, τον τραπεζικό κλάδο. Και Προφανώς δεν θα εξαρτάται η δουλειά τους από το ποια τράπεζα ε, έχει πρόβλημα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την, το ρυθμό, τους ρυθμούς μας όσον αφορά την προπαρασκευαστικές, τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Θα πρέπει να δώσουμε τα σωστά μηνύματα από την αρχή έτσι ώστε να είναι ο τραπεζικός κλάδος ασφαλής και ε, έχει γίνει ε, μια προσπάθεια αξιολόγησης ε, πρόσφατα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο τελευταίο Συμβούλιο της ΕΚΟΦΗΝΑ, αποφάσισε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας τα τελευταία στοιχεία για την αξιολόγηση. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είμαστε υπόλογοι και ε, πραγματικά θέλουμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είμαι, θέλω να ε, ασκήσω τα καθήκοντά μου σεβόμενοι το πνεύμα και το γράμμα της Διαθεσμικής Συμφωνίας έτσι ώστε να έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το γεγονός αυτό το ότι είμαι υπόλογη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει και την δύναμη των ελεγκτών Επίση, ε, Επίσης, ε, μια άλλη πρόκληση είναι να υπάρχει μια επικοδομητική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο προσωπικό, ε, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο ε, η επιτυχία του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας εξαρτάται από την ε, καλή συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα συστατικά του στοιχεία, κυρίως ανάμεσα στις εποπτικές, στις εποπτικές ομάδες που εξασφαλίζουν την εποπτεία 160 σημαντικών τραπεζών. Πέραν τώρα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, το να πετύχουμε την ολοκλήρωση του ενός εποπτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο είναι ε, ύψης της σημασίας. Αυτή η ολοκλήρωση ε, ε, θα λαμβάνει υπόψη και την δράση της ΕΜΠΑ και θα πρέπει να, να προσέξουμε ιδιαίτερα τον ρόλο ε, της, ε, του ενιαίου αποπτικού μηχανισμού στα θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την φωνή της Ευρώπης σε διεθνά φόρα. Ε, η, τελευταία πρόκληση είναι ότι θα πρέπει ε, σε, σε χρόνο να ενισχύσουμε ε, τους πυλώνες τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο παίζουν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τους όρους του Κοινοβουλίου. Για να τα πούμε τα πράγματα απλά, πιστεύω ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δεν θα δώσει όλα του τα... δεν θα δώσει τα αποτελέσματα που περιμένουμε, εάν δεν είναι ε, ε, ρωμαλαίος αν θέλετε και εάν δεν ολοκληρωθεί ο τρίτος πυλώνας. Κυρία Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και είμαι έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. θα χρονομετρήσω τις, το χρόνο των ε, ερωτήσεων. Υπάρχει ήδη ο κατάλογος ε, των ομιλητών. Ε, δεν χρειάζεται τώρα να, μου, να κουνάτε τίποτα από τα χέρια σας. Πρέπει να είστε ήδη στο κατάλογο. Ζων Πόλ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Νουή, σας επέλεξε το Συμβούλιο των ε, Διοικητών των Τραπεζών για να ε, είστε υποψήφια. Ε, περάσατε ήδη ένα εμπόδιο, το, την ιδιωτική ακρόαση και δεν πρόκειται να είμαι πρωτότυπος. Θα ακολουθήσω την ίδια σειρά, των, το ίδιο πνεύμα των ερωτήσεων που έγινε εκεί στην ιδιωτική ακρόαση. Ε, ήσασταν ε, από τους υποψηφίους που επελέγησαν στο τέλος και που ε, πληρείται τα περισσότερα προσόντα από αυτά τα οποία απαιτούνται ε, και δημοσιεύθηκαν στις 29 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Απάντηση. Πιστεύω ότι η ανάγκη να έχουμε μια μεγάλη εμπειρία, αν θέλετε, μια μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα του ελέγχου και της εποπτείας είναι ένα σημείο κλειδί και μπορούμε να, μπορεί να μπορούμε να δούμε ότι δεν έχω εμπειρία σαν τραπεζίτης ή τραπεζικός, το οποίο θα ήταν ένα ατού βέβαια. Αλλά τέλος πάντων όλες οι αποστολές αν θέλετε ε, εποπτείας ή ελέγχου και σε περίοδο κρίσης κυρίως είναι ένα πλεονέκτημα. Επίσης ε, θεωρώ ότι η επιτυχία της ε, λειτουργίας ε, της, ελεκτρικής αρχής των τραπεζών στην Γαλλία είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα και το θέμα αυτό ήταν δύσκολο γιατί οι, επόπτες αν θέλετε των ασφαλιστικών εταιριών δεν αντιμετώπισαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την προπτική αυτή να υπάρξει δηλαδή μια ελεκτρική αρχή αλλά οι ικανότητές μου κατάφεραν έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλοι να συνεργαστούν σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης, διαφάνειας και ε, εποφεληθήκαμε από τα προσόντα και τις ικανότητες των μεν και των δε και πιστεύω ότι η διεθνής εμπειρία και η ευρωπαϊκή εμπειρία που είχα ούτως ή άλλως στο παρελθόν θεωρήθηκε αρκετά σημαντική. Ούτως ή άλλως πάντοτε ε, ήμουνα εθελόντρια αν θέλετε, λόγω ενθουσιασμού και λόγω πάθους αν θέλετε, ε, για να ε, ολοκληρωθεί, για να δημιουργηθεί μάλλον η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και όταν ήμουνα στη Βασιλεία το 2003, μόλις είχε δημιουργηθεί το ΣΕΠΣ, και ο συνάδελφος, ο κύριος Χοϊντάν, ήταν, είχε επιλεγεί σαν πρόεδρος. Αν περιμένουμε Υπάρχει και αντιπρόεδρος, αλλά τέλος πάντων ούτω ή άλλω ε, είμαι υποψήφια για πρόεδρος. υπήρχαν και άλλοι υποψήφοι, αλλά τέλος πάντων ε, ε, τα πράγματα προχώρησαν. πάντοτε ήθελα να είμαι πρόεδρος διαφόρων ομάδων, πάντοτε στη δουλειά μου έδειχνα και πάθος και ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι και η εμπειρία που απέκτησα στη Γαλλία και ενώπιον του Γαλλικού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Οικονομικών και της Γερουσίας και της Βουλής, η ικανότητα να αντιμετωπίζω ακροάσεις σαν και αυτή την σημερινή, δείχνει ακριβώς ότι κάνουμε και στον τομέα της εποπτείας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πολύ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ελίσσα. <laughs> I was, already... Ήμουν έτοιμη να δώσω το λόγο στον Άντζελη, αλλά έχετε δίκιο. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που είστε μεταξύ ημών. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Η έναρξη των, λειτουργών, των λειτουργιών ε, εποπτείας μέσω του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού SSM είναι ένα από τα σημεία κλειδιά της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Νομίζω ότι οι πολίτες θα ήθελαν να γνωρίζουν πώς με βάση όλη σας την πείρα θα αντιμετωπίσετε το συντονισμό των εθνικών μηχανισμών εποπτείας όταν πρόκειται για τράπεζες πολύ πιο ε, μικρής εμβέλειας. Πώς θα εντάξετε λοιπόν την επιτήρηση αυτών των τραπεζών στο γενικότερο πλαίσιο. Δεν είναι εύκολο να επιτύχει κανείς τη χρυσή τομή γιατί οι καταστάσεις ε, στις χώρες μέλη είναι τόσο διαφορετικές. Δεύτερον, θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε ούτω ώστε να έχουμε μια επιτήρηση και εξυγίανση με τόσο διαφορετικούς κανόνες που υπάρχουν ή θεωρείτε ότι θα προχωρήσουμε ούτω ώστε η εποπτεία και η εξυγίανση να γίνονται με ενιαίο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την ε, ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων. Τρίτον, η σχέση μεταξύ της εποπτείας εντός της Τραπεζικής Ένωσης και εκτός της Τραπεζικής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε εγγυήσεις ότι το ότι εντός της Τραπεζικής Ένωσης θα έχουμε πιο ισχυρή εποπτεία δεν θα δημιουργήσει ανισορροπίες στην εσωτερική αγορά. Θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας και για αυτό το θέμα. Γιατί σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, την ΕΜΠΑ. Όσον αφορά την εργασία που από κοινού που θα πρέπει να γίνει με τις εθνικές ε, αρχές, τις εθνικές τράπεζες. Νομίζω ότι ήδη ε, στελεχωνόμεθα, έχουμε ήδη αρχίσει να προσλαμβάνουμε προσωπικό, έχουμε λάβει θαυμάσιες αιτήσει από διακεκριμένα άτομα που έχουν ε, ευρωπαϊκή προοπτική θεωρούν ότι το SSM είναι πολύ σημαντική, μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη για να βελτιωθεί η ποιότητα της εποπτείας στην Ευρώπη. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, το κατάλληλο κλίμα για να δράσουμε υπέρ του ευρωπαϊκού συμφέροντος γενικά. Ήδη έχουμε αρχίσει να καταγράφουμε το οργανόγραμμα. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε κοινέ ομάδες εποπτείας. Για παράδειγμα, θα υπάρχει ένα συντονιστή σε κάθε μία τέτοια ομάδα κοινή εποπτείας ε, και αυτοί θα είναι, οι υπόλοιποι θα είναι 5, 6 ή 10 για να ε, εποπτεύουν την Deutsche Bank για παράδειγμα Ορισμένοι θα είναι στη Φραγκφούρτη, αλλά θα έχουν ανταποκριτέ και στι άλλε χώρε όπου υπάρχουν παραρτήματα τη Deutsche Bank. Αυτέ είναι καλέ ιδέε επιπλέον. Η θέση αυτή για την οποία είμαι υποψήφια είναι η πιο ενδιαφέρουσα και πιο απαιτητική από πλευρά διοίκηση να διοικούμε ομάδες που υπάγονται σε διαφορετικές αρχές, σε διαφορετικές χώρες. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν αυτές, όχι μόνο, θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν και σε αυτό αναφερόμουν, τους επικεφαλείς αυτών των, ε, αυτών των κοινών ομάδων. Λοιπόν, από τη μία έχουμε το δικό μου μηχανισμό και από την άλλη έχουμε το μηχανισμό για την εξυγεία των τραπεζών, SRM. Γι' αυτό υπάρχουν δύο διαφορετικές αρχές. Αλλά νομίζω ότι ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, SRM, πρέπει να αφορά όλες τις τράπεζες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Περιφέρειας. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο οι πιο σημαντικές μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά εάν τελικά καταλήξουμε σε αυτό, δεν θα είναι η βέλτιστη λύση. Καλύτερα να συμπεριλαμβάνονται όλοι. Όσον αφορά το ρόλο που θα παίξει ο SSM με την ενία αγορά, δηλαδή σχέσεις με την EBA, νομίζουμε ότι ο SSM είναι ατού για την ε, EBA, γιατί θα εγγυηθεί ότι θα υπάρχει συνεπής αντιμετώπιση. Χρειαζόμαστε την ε, EBA, την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η επικεφαλής της EBA, ε, ο επικεφαλής της EBA και εγώ γνωριζόμαστε πολύ καλά, ήμασταν στα ίδια όργανα και ε, μ' αρέσει πολύ η συνεργασία και πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλά και η EBA είναι επίσης ατού για τον SSM γιατί έχουμε το ενιαίο βιβλίο κανόνων, το ενιαίο βιβλίο ε, εποπτείας έχουμε δεσμευτικά κριτήρια, δεσμευτικές προδιαγραφές ε, για το βαθμό έκθεσης των τραπεζών. Θα έχουμε λοιπόν πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούμε με την EBA τα επόμενα χρόνια. Με συγχωρείτε που ήδη είπα πολλά, αλλά ε, έχω ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και στις γραπτές απαντήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Αλντέι Σιλβί ευχαριστούμε και <clears throat> είμαι ιδιαίτερος ευτυχή που παρευρίσκεστε. Θα ήθελα να σας ε, θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τις διεθνείς προοπτικές. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι θα επιδιώξουμε την ε, ένταξη αυτού του εποπτικού μηχανισμού στην ε, στον κόσμο παγκοσμίω, στη διεθνή σκηνή και θα έλεγα ότι συχνά στην Ευρώπη εστιάζουμε περισσότερο στα εσωτερικά μας, στα ευρωπαϊκά θέματα. Εσείς έχετε μια διεθνή εμπειρία, έχετε ε, δουλέψει στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ε, βλέπετε αυτή τις συνεργασίες πέρα από διπλωματικές σχέσεις και φιλικές σχέσεις ε, Πώς μπορούμε, για παράδειγμα, σε μια παγκόσμια αγορά όπου οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ε, στην Αμερική, στην Ασία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, να τοποθετηθούμε εμείς όταν συχνά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε άλλα κέντρα. Πιστεύω ότι η φωνή της Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει, να ακουστεί και χρειάζεται να υπάρχει μια συνοχή, δηλαδή να εκφραζόμαστε με μια φωνή. Δυστυχώς αυτό δεν σημαίνει πάντα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την άποψή της στα διεθνή φόρα και ε, ευελπιστώ ότι η δημιουργία του SSM θα βελτιώσει την κατάσταση. Ε, χρειάζεται επίσης συντονισμός με την EBA, μιας και πρόκειται και οι δύο αυτοί οργανισμοί να παρίστανται σε διεθνείς συναντήσεις. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι πρέπει να μην ξεχνάμε τις, διάφορε, τις διαφορετικότητες, τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ε, χρηματοπιστωτικών αγορών στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Δηλαδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην ευρωπαϊκή αγορά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το 75% ε, των χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών είναι, γίνεται από τις τράπεζες είναι κάτι που μας ξεχωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε. Χρειάζεται λοιπόν μια νομοθετική πρωτοβουλία όσον αφορά τη δομή των τραπεζών στην Ευρώπη και το ζήτημα της ε, διάκρισης. Ε, ε, έχουν αναλυθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στη Γαλλία, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό. Και σκοπεύω να δραστηριοποιηθεί ο SSM σε αυτόν τον τομέα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την δομή της χρηματοδότησης της οικονομίας στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε με τις λεγόμενες ενέργειες market making, δηλαδή την χρηματοδότηση επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Θα χρειαστεί λοιπόν να βρούμε λύσεις γραμμένα στα μέτρα της Ευρώπης. και σίγουρα θα συνεργαστούμε με το ε, επαρκές προσωπικό που προσλαμβάνουμε έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιωτερότητες της Ευρώπης στις πολιτικές που θα εφαρμόσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε για τους πράσινους. Φεν. Καλώς ήρθατε. Δύο ερωτήσεις κατά βάση η πρώτη. Όπως θα γνωρίζετε πριν την σημερινή μας ακρόαση, διεξήχθη μια μεγάλη διαπραγμάτευση, ορισμένες φορές επίπονη, σε σχέση με την σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτόν τον εφορέα. Δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί τις εργασίες σας και υποβάλαμε μια σειρά ερωτημάτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δυστυχώς, οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ασαφείς, παρά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις μας ήταν σαφές. Για παράδειγμα, ρωτήσαμε ποια ήταν τα μέλη των προπαρασκευαστικών ομάδων για τη δημιουργία του SSM. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα ονόματα τους και το οργανόγραμμα του οργανισμού στο μέλλον και δεν τα λάβαμε αυτά τα στοιχεία. Ρωτώ λοιπόν, δεσμεύεστε να απαντήσετε Πλήρω σε αυτές τις ερωτήσεις. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητα τα οποία σεβόμαστε, αλλά πέραν αυτού δεσμεύεστε να απαντήσετε πλήρως τα ερωτήματα που έχουμε θέσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί πράγματι μια ε, σχέση αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του διαχωρισμού, τη παρακολούθηση και τη υποπτία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι αυτές οι κρίσιμες λειτουργίες θα διαχωριστούν. Για παράδειγμα, το τομέα ανθρωπίνων πόρων ή ο τομέα διεθνών σχέσεων ή το τομέα νομικών υπηρεσιών θα είναι ξεχωριστή για τους μεν και τους δε. Προσωπικά πιστεύω ότι οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου στα θέματα διαφάνειας αλλά και ε, του, ότι πρέπει να είμαι θα υπόλογια του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικά και ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες υποφέρουν από την κρίση σήμερα και αυτή η κρίση προκλήθηκε από τον, ε, από τον δημοσιονομικό τομέα και είναι απέτηση των πολιτών να ξέρουν τι κάνουμε και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί και θα πρέπει να προσφέρουμε πληροφορίες ε, στους εκπροσώπους των πολιτών. Αυτό είναι μέρος των καθηκόντων μου. Ε, όπως σας είπα, είμαι ε, αποφασισμένη πλήρως να σεβαστώ το πνεύμα και το γράμμα των διεθνισμικών συμφωνιών. Πρέπει να σας πω ότι είμαι συνηθισμένη σε κάτι τέτοιο Έχω μελετήσει πολύ προσεκτικά το περιεχόμενο των συμφωνιών, της συμφωνίας και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην το έχω κάνει ήδη ε, και στις ακροάσεις ε, στο, στην, Γαλλική Βουλή και στην Γερουσία. Είναι ένα κομμάτι των ε, καθηκόντων μου, των, καθηκόντων, των σημερινών μου καθηκόντων. Δεν υπάρχει πρόβλημα επομένως. Προσπαθώ να απαντήσω στην ερώτησή σας, ίσως να μακρηγόρησα λίγο στις απαντήσεις μου, αλλά ε, αποφάσισα να στείλω τις απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις ε, πριν την ακρόαση. Όχι, όχι, δεν ασκούσα κριτική, απλώς οι, ε, εκείνες οι ερωτήσεις ήταν κάπως ελλειπείς. Κοιτάξτε, το μόνο, η μόνη λεπτομέρεια που θα μπορούσα ίσως κάπως να διαφοροποιήσω ε, είναι να πω ότι ε, εργάζομαι σε μια κεντρική τράπεζα που ασχολείται και με τα θέματα εποπτείας και είμαι υπεύθυνη με, την, ε, με τα θέματα διεύθυνσης της τράπεζας. Ξέρω ποιες είναι οι αρχές. Ξέρω ότι υπάρχει διαφορετική γραμμή, αν θέλετε, όσον αφορά ε, την, ε, τον, ε, και τις δύο αυτές δραστηριότητες. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για μένα, απλώς μία απόχρωση αν θέλετε. Όσον αφορά την εσωτερική κινητικότητα του προσωπικού, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα ανάμεσα στο εποπτικό και μη εποπτικό κομμάτι της τράπεζας στη Γαλλία και αυτό είναι ένα ε, ε, κριτήριο, αν θέλετε, ένα πλεονέκτημα για να προσελκύσουμε κόσμο. Διότι πολλοί δεν θέλουν να μείνουν σε ένα συγκεκριμένο ε, τομέα, σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, α πούμε, την εποπτική και θέλουν στη διάρκεια της καριέρα του να μετακινηθούν. Θέλουμε να έχουμε ούτως ή άλλως ένα, μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή και ένα ανεξάρτητο κανάλι, αν θέλετε, για το πώς θα διευθυνθούν οι πληροφορίες που αφορούν ε, το εποπτικό κομμάτι. Ικανοποιηθήκατε? στο διεθνές ε, νομικό, σε επίπεδο ε, ε, διεθνούς νομικού επίπεδου, ε, τμήματος, συγγνώμη, τι θα γίνει. Ναι, όντως θα υπάρχει μια διεθνής μονάδα σε οριζόντιο επίπεδο που θα έχει πολλές λειτουργίες, διεθνές τμήμα για την εποπτεία και θα υπάρξουν, θα, θα, θα στελεχωθεί με δικηγόρους, με νομικούς, Ακόμα συζητάμε με την ECB, με την έκτο τέλος πάντων, ε, πώς θα οργανωθεί η γραμματεία της, ε, του ενιαίου μηχανισμού, γιατί και εκεί πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι νομικοί, διότι τα άτομα αυτά θα είναι οι τελευταίοι αν θέλετε που θα εξετάζουν τις σημειώσεις, ε, τα έγγραφα ε, των εποπτών, των ελεγκτών και θα πρέπει κάποιος να ελέγχει ότι είναι γραμμένα όλα αυτά στη σωστή νομική γλώσσα. και θα πρέπει να ε, συντάσσουμε εκθέσεις σε τρεις κατηγορίες ε, νόμου, αν θέλετε, σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, την που προέρχεται από τις συνθήκες, αυτό είναι εύκολο, ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα προέρχεται από τις οδηγίες και εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο μετατίθεται οι, μετατίθεται οι ευρωπαϊκές οδηγίες σε εθνικό δίκαιο. Μετά θα υπάρχουν και οι εκθέσεις με βάση την εθνική νομοθεσία. Άρα χρειαζόμαστε νομικούς οι οποίοι να είναι απόλυτα καταρτισμένοι και να μπορούν να στελεχώσουν ε, ε, τον κανονισμό, τον μηχανισμό, συγγνώμη. Ο κύριος κυρία Νουή, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Είπατε κατά την παρουσίαση των ε, απόψεών σας, το ξέρουμε, ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού είναι να ελέξει αυστηρά τα στοιχεία των ενεργητικών των μεγαλύτερων τουλάχιστον ευρωπαϊκών τραπεζών και να ολοκληρώσει τα νέα stress test. Βασική επιδίωξη αυτού του ελέγχου είναι να εξακριβωθεί αν υπάρχει η απαραίτητη κεφαλαϊκή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών που έχει τεθεί στο όριο του 8%. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξή παράδοξο και εκεί θα εστιαστεί η ερώτησή μου. Με βάση το ελληνικό μνημόνιο, με βάση το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας για τις ελληνικές τράπεζες για την διετία 2012-2014 έχει τεθεί στο 9% και όχι στο 8%. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε κυρία Νουή δημιουργεί πρώτον ανισότιμη μεταχείριση μεταξύ των τραπεζών σε μια περίοδο που οι ελληνικέ τράπεζε έχουν αναδιαρθρωθεί με εξαγορές, συγχωνεύσεις και Και δεύτερο, έχει επιπτώσει στην πραγματική οικονομία, καθώ δύο δισεκατομμύρια δεσμεύονται από αυτόν τον περιορισμό που σα ανέφερα και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρέ μεσέ μεγάλε επιχείρησει που όπω ξέρετε στην Ελλάδα κλείνουν. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξή: ω πρόεδρο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού σκέφτεστε να εισηγηθείτε να μειωθεί αυτός, αυτό το όριο για τις ελληνικές τράπεζες ούτως ώστε να εναρμονιστεί με τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή το 8%. Σας ευχαριστώ πολύ. I am sorry to respond that uh, I cannot uh, take... Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να δεσμευτώ προς αυτή την κατεύθυνση. Αν με επιλέξετε θα είμαι απλώς πρόεδρος ε, του SSM του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού. Οπότε, υπ' αυτήν μου την ιδιότητα, θα πρέπει να είμαι σίγουρη ότι η αποτίμηση του ισολογισμού στα πλαίσια των stress test θα γίνει με αυστηρή μεθοδολογία, με ομάδες που θα έχουν κεντρική καθοδήγηση, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε, στη θέση του οδηγού, με την συνεργασία και άλλων επιτηρητικών αρχών, με σωστή διακυβέρνηση, σωστή συνεργασία με τους εθνικούς επιτηρητές με, μέσω και της μόνιμης επιτροπής ε, των πραγματικών ισολογισμών και διασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλα αυτά τα επίπεδα. Αυτή είναι η εντολή μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Ανάλογα τώρα από την κατάσταση των τραπεζών. Ανάλογα με την κατάσταση των τραπεζών μια χώρα ή μια τράπεζα συγκεκριμένα, οι αρχές επιτήρησης, αρχές εποπτείας έχουν τα ενηγκαία μέσα, τα αποκαλούμε εργαλεία ε, πιλοταρίσματος για να ζητήσουν να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα για κάποια τράπεζα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για το αν είναι υπερβολικό αυτό που απαιτείται ή όχι, αλλά θα ήθελα να έχετε υπόψη ότι δεν είναι μόνο οι ελληνικές τράπεζες από τις οποίες ε, απαιτείται αυτό το 9%. Με το πρόγραμμα Pilot 2 το ζητάω και από ορισμένες γαλλικές τράπεζες. Άρα δεν υπάρχει θέμα ότι υφίστανται διακρίσεις οι ελληνικές τράπεζες, επειδή είναι ελληνικές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και πάλι το ΕΛΚ. Η Νοριάν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας χαίρω για την επιλογή σας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ήθελα να σας κάνω τις εξής ερωτήσεις. Η κυρία Λαγκάρντα κάποτε είπε ότι ότι αν ε, η τράπεζα λεγόταν Lehman Sisters και όχι Lehman Brothers, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικό σήμερα. Δηλαδή οι γυναίκες αντιμετωπίζουν και διαχειρίζονται καταστάσεις κινδύνου διαφορετικά από τους άνδρες. Είναι πιο προσεκτικές, πιο επιφυλακτικέ. Εάν ε, θεωρήσουμε ότι ισχύει αυτό που είπε η κυρία Λαγκάρντ, ε, θα πρέπει να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική ισότητα φίλων για το, στον τομέα αυτό δεν είναι δευτερεύον θέμα. Το έχουμε συζητήσει ε, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανειλημμένα. Και το ερώτημά μου είναι τι θα κάνετε για να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει αρκετή εκπροσώπηση και των δύο φίλων στο νέο αυτό SSM. Και το άλλο που ε, απορρέει από συζητήσεις που κάναμε κατά τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό του SSM, πώς βλέπετε τη σχέση μεταξύ ε, των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του SSM στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, αυτές οι δύο λειτουργίες ε, ήταν εναλλάξιμες σε ένα βαθμό. Και εμείς ε, θεωρούμε ότι ο πρόεδρος που εξορισμού δεν είναι μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να είναι ο επικεφαλής και ο αντιπρόεδρος που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ θα πρέπει να παίξει το ρόλο αντιπροέδρου και το πολύ να μπορεί να υποκαταστήσει, το, το μπορεί να μπορεί να εκπροσωπήσει τον πρόεδρο. Και έχετε δίκιο ε, για αυτά που είπατε για τον μηχανισμό εξυγίανση των τραπεζών. Αλλά η απάντησή σας ε, νομίζω ότι χρειάζεται να διευκρινιστεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι υποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ε, ε, ζητήσουν τη δημιουργία του μηχανισμού αυτόνομα. Θα ήθελα να άποψή Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να εργάζομαι σε περιβάλλοντα που, όπου υπάρχει διαφορετικότητα. Έχω εργαστεί σε 15 μελές σώμα με 13 διαφορετικές εθνικότητες. Πολύ ενδιαφέρον ε, περιβάλλον και το φύλλο δεν είναι το μόνο κριτήριο, αλλά είναι και αυτό ένα από τα κριτήρια της διαφορετικότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να προωθήσουμε, να ευνοήσουμε καλύτερα τις γυναίκες στον ε, μηχανισμό εποπτείας. Έχω συναδέλφους από τη Γερμανία, από τη Φιλανδία, γυναίκες και είναι πολύ καλές στη δουλειά τους, ε, εκτιμώνται από όλους. Κατά τη γνώμη μου, στον τομέα τον εποπτικό, οι γυναίκες θα πάνε μια χαρά. Ωστόσο, ωστόσο, θεωρώ ότι η πρόσληψη προσωπικού στον SSM πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα αξιοκρατική. Χρειαζόμαστε άτομα που να έχουν τις αναγκαίες ικανότητες, που να είναι διατεθειμένοι να μάθουν ακόμη περισσότερα, να εργαστούν σκληρά, να εργαστούν σκληρά για να μάθουν ακόμη περισσότερα. Είναι δύσκολο να βρούμε τέτοια άτομα. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρούμε και γυναίκες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα και φυσικά και των φίλων. Αλλά πρέπει η βάση μας να είναι η αξιοκρατία για τις προσλήψεις. Τώρα για το ρόλο Προέδρου-Αντιπροέδρου. Αυτά που υπόθηκαν για Lehman Brothers και Lehman Sisters. Το πιο σημαντικό δεν είναι ποιος είναι ο αρχηγός. Το σημαντικό είναι η καλή διακυβέρνηση. Όταν είσαι πρόεδρος πρέπει να είσαι ο αρχηγός. Ανεξαρτήτως φίλου. Και όλοι πρέπει να το καταλαβαίνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι επικεφαλής ενός οργανισμού με 1.100 υπαλλήλου και διορίστηκα ακριβώ από την κυρία Λαγκάρντ που θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάποιον άλλον μετά τη συγχώνευση. Προηγουμένω δικούσα ένα οργανισμό 600, τώρα 1.100. Αλλά πιστεύω ότι αν είχε την παραμικρή αμφιβολία για τι ε, ηγετικέ μου ικανότητε για να δικήσω ένα τέτοιο μηχανισμό, δεν θα με είχε διορίσει. Όσον αφορά ποιος μπορεί να προκαλέσει τη διαδικασία εξυγίανσης μιας τράπεζας. Αυτή ήταν η ερώτησή σας. Ε, ίσως να μην ήταν τόσο σαφής η απάντησή μου γιατί έχω και εγώ κάποιες αμφιβολίες. Η εποπτική αρχή είναι στην καλύτερη θέση για να δει αν έχει προβλήματα μια τράπεζα, αν θα πρέπει να μπει στη διαδικασία εξυγίανσης, αν θα πρέπει να είναι μόνος εποπτικός μηχανισμός για να προκαλέσει την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης. Η απάντησή μου είναι ίσως όχι. Νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο πρόεδρος ε, της υποπτικής αρχής να ρωτήσει εάν θα πρέπει να υπάρξει ε, εξυγίανση. Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές χώρες. Και αυτό ίσως επειδή είναι τόσο ευαίσθητο θέμα και δεν υπάρχει ε, μία απάντηση για όλες τις περιπτώσεις. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν αρκετά συγκεκριμένη και σε αυτή τη δεύτερη απάντηση. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να παίζει ε, πολύ ισχυρό ρόλο ο πρόεδρος του SSM, αλλά θα πρέπει να είναι ο μόνος που να ξεκινάει την εξυγένση. Δεν είμαι σίγουροι γι' αυτό. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να πω περισσότερα σήμερα για το θέμα αυτό. Έχω την ε, αίσθηση ότι και άλλοι θα έπρεπε να έχουν ένα ρόλο όχι οι άλλοι να παίζουν το ρόλο της πρόκλησης, αλλά να παίζουν ρόλο στην πρόκληση. Ναι, ε, το θέμα είναι ποιοι άλλοι θα έπρεπε να παίζουν ρόλο σε αυτή την πρόκληση εξυγίανσης. Και εδώ είναι και το πρόβλημα. Ελκ και πάλι. Μπένχαρντ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. κύρια Νουή, χαίρομαι που είστε εδώ στο Κοινοβούλιο για αυτή την ακρόαση. Δύο ερωτήσεις. Δύο μάλλον ε, κύκλους θεμάτων που θέλω να κάνω ερωτήσεις. Πρώτον, τα κρατικά ομόλογα. Κατά της ε, πρότασης που έγινε, ε, ο κύριος Ντράγκη δεν ακολούθησε αυτή τη σύσταση και ο κύριος Ντράγκη επανέφερε το θέμα σε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Για μένα ο πρόεδρος ε, της ε, ΕΚΤΑΦ δεν θα είχε καμία, ε, κανένα συμφέρον να προκαλέσει ανησυχίες στις αγορές για αυτά τα κρατικά ομόλογα. Ως επικεφαλής του ενιαίου μηχανισμού θα πρέπει να ενδιαφέρεστε για το πώς θα καλύψετε τους ισολογισμούς, να μειώσετε τα ελλείμματα των τραπεζών. Γι' αυτό προσωπικά Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της εκτίμησης του κινδύνου για τα κρατικά ομόλογα, τώρα που έχουμε και αυτά, αυτήν την επικείμενη ε, διαδικασία ελέγχου των ισολογισμών των τραπεζών και εάν υπάρξουν ε, στο μέλλον τέτοιες ε, συγκρούσεις απόψεων με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πώς θα το αντιμετωπίσετε. Το άλλο το ανέφερε και η συνάδελφος Φεραίρα, αλλά θέλω να ρωτήσω ακόμη περισσότερα τι δυνατότητες και μεθόδους βλέπετε, ούτως ώστε στην πράξη η εποπτεία να λαμβάνει υπόψη το μικρό βαθμό πολυπλοκότητας μικροτέρων τραπεζών συγκεκριμένα. Θεωρείται ότι θα έπρεπε να διατηρηθούν οι εθνικές αδειότητες εποπτείας για μικρότερες τράπεζες. Άλλη ερώτηση. Τι άποψη έχετε για τη χρήση της γλώσσας της χώρας στην ε, ε, επικοινωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών μιας συγκεκριμένης χώρας. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τον κρατικό δανεισμό και την ε, έκθεση του δημοσίου χρέους, γίνονται πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι η στιγμή βέβαια να κάνουμε σκηνές δραματικές ε, δημόσια για αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχουν κανόνες. Ε, καταρχάς ε, στην αξιολόγηση των ισολογισμών στα τρέστ τεστ, η ΕΜΠΑ πέρυσι είχε προσφέρει συγκεκριμένους κανόνες και κριτήρια και τρόπο ελέγχου αν θέλετε και αξιολόγησης της έκθεσης των τραπεζών. Οτιδήποτε όμως και να κάνουμε, η κεφαλαιακή ε, επάρκεια ε, δεν θα είναι ποτέ αρκετή. Ε, ένα σημαντικό εργαλείο είναι να περιορίσουμε τις μεγάλες εκθέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην έκθεση από ό,τι, καταλα... από ξέρω υπάρχουν επόπτες που ήδη ε, περιορίζουν τις μεγάλες εκθέσεις και εκθέσεις ε, σε όλα τα και δημόσια, ε, σε δημόσιο χρέος και σε ιδιωτικό χρέος. Και το απαιτούν αυτό διότι θεωρούν ότι είναι ένα στοιχείο επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου. Αυτό το οποίο κάνουμε επίσης και στην αξιολόγηση των ισολογισμών είναι να δούμε ποια είναι τα πιο ε, ε, παρακινδυνευμένα αν θέλετε χαρτοφυλάκια και για το δημόσιο χρέος ούτως ή άλλως αλλά και για το μέσα στα πλαίσια του, στον stress test έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να δούμε και να ελέγξουμε το δημόσιο χρέος. Και Νομίζω ότι υπάρχουν, ε, πρέπει να εφαρμόσουμε και κανονισμούς ε, και στα θέματα ρευστότητας ε, που είναι ένα κίνητρο να περιορίσουμε τον, την έκθεση στο δημόσιο χρέος. διότι εάν έχουν ε, ε, ένα μεγάλο μερίδιο στο δημόσιο χρέος δεν θα μπορέσουν να ε, κάνουν καλά τη λειτουργία τους. Επίσης η ερώτησή σας αν κατάλαβα καλά έχει να κάνει με το σύστημα εξυγίανσης των τραπεζών το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλες τις τράπεζες ή μόνο για τις σημαντικές τράπεζες. Πιστεύω ότι είναι εφικτό Ίσως ε, είναι καλύτερο το να έχουμε μία ενιαία αρχή για όλες τις τράπεζες. Έχω την εντύπωση ότι είναι εφικτό βέβαια ε, για τις μεγαλύτερες τράπεζες που έχουν ε, τις, τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρογνωμοσύνη, που έχουν ήδη έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν την εξυγίανση. Εάν μπορεί να ε, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα του opt-out για τις χώρες που μπορούν να το κάνουν από μόνες τους. Αλλά επειδή όμως ε, έχω ένα ευρωπαϊκό, έχω ένα ευρωπαϊκό προστατολισμό, ε, πιστεύω ότι είναι καλύτερο ένα ενιαίο σύστημα αντιμετώπισης. Ανέφερα και το θέμα αν είναι δυνατόν στην επικοινωνία μεταξύ των τραπεζών μιας χώρας και της Γρήσης Τράπεζας να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της χώρας. Κοιτάξτε, επειδή μεγαλύτερα ξέρετε πόσο σοβαρό αυτό το θέμα η χρήση της γλώσσας της χώρας. Οπωσδήποτε θα σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όλες οι εποπτικές αρχές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ενημέρωση στα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ελληνικά ή άλλες εθνικές γλώσσες. Και ο SSM θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας. Ολοκληρώνουμε τώρα ένα πλαίσιο λειτουργικό, νομικό, εφαρμογής του κανονισμού για τον SSM θα διανεμηθεί, θα υπάρξει διαβούλευση και έτσι θα δείτε ότι αυτά οπωσδήποτε θα τα σεβαστούμε και είναι πολύ σημαντικά. Ωραία. Από τους ελστές Αντολίν. Ευχαριστώ και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις και μετά την ιδιωτική ακρόαση. Πρώτον, σας ευχαριστώ που εκφράσατε δέσμευση να εφαρμόσετε τις συμφωνίες με το Κοινοβούλιο από πλευράς Δημοκρατικού Ελέγχου και στο πνεύμα και στο γράμμα. Να είναι σαφές ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ούτε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψεις όχι μόνο με τον πρόεδρο, την πρόεδρο του SSM, αλλά και με τα ε, πιο σημαντικά μέλη, όπως ακριβώς τα προβλέπει το, ε, η Διοργανική Συμφωνία για να υπάρχει πραγματική δημοκρατική λογοδοσία. Δεύτερον, με αυτά που είπε ένας συνάδελφος για τον κίνδυνο από τα κρατικά ομόλογα, το δημόσιο χρέος. Εγώ είδα δύο δημοσιεύσεις. Μία που αναφέρεται τα τελευταία δύο χρόνια οι επιπτώσεις της εποπτείας και αν το αντιμετωπίζει σωστά ε, ο ρυθμιστικός μηχανισμός του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή να αποφύγουμε τις ε, ανεπιθύμητες επιπτώσεις από αυτή την έκθεση. Η δημιουργία του ΣΣΜ είναι άλλο ένα βήμα στην ενδυνάμωση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια συνοχή με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει. Να δημιουργήσουμε δηλαδή διαφορετικέ κατευθύνσει από αυτήν που για παράδειγμα ε, περιλαμβάνεται στο μνημόνιο για την Ισπανία. Δεν θα ήταν ε, λογικό κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρχει συνοχή και να καταλάβουμε ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να βοηθήσουν να μειώνεται η ένταση επί του δημοσίου χρέους και να δημιουργηθεί πάλι η δυνατότητα δανειοδότησης. Δηλαδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι σε πιο ρωμαλαία κατάσταση. Ευχαριστώ όσον αφορά την διοργανική συμφωνία. Είναι δεδομένη η δεσμευσή μου να την τηρήσω και ως προς το γράμμα, ως προς και το πνεύμα. Τώρα θα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα σας ε, επισκέπτομαι πιο τακτικά και περισσότερο και το προτιμώ αυτό, γιατί έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να υπάρχει διαφάνεια στις επικοινωνίες μεταξύ μας. Όταν είναι ε, αραιές οι συναντήσεις μας, ε, αναγκαστικά θα μου ζητάτε να, να παράσχω πληροφορίες μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά και δεν είναι αυτό στις προθέσεις μου. Είναι καλύτερα να έχουμε τακτικές συχνές ε, συναντήσεις και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και όταν υπάρχουν προβλήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια μακροχρόνια σχέση ε, εμπιστοσύνης. Όσον αφορά τα κρατικά, το κρατικό χρέος και τις ε, ανεπιθύμητες επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η εποπτεία τον τομέα αυτών, πράγματι αυτή τη στιγμή υιοθετούνται διάφοροι νέοι κανονισμοί, ε, η 2, το CDR περισσότερα και νέα stress test, τα οποία ε, εστιάζουν περισσότερο στον, ε, στο κρατικό χρέος και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα νέα τεστ δεν θα δημιουργήσουν περισσότερες δυσκολίες από τις ήδη φυστάμενες. Άρα πράγματι, θα λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση που δημιούργησε το μνημόνιο. Πρέπει να πω ότι στη χώρα μου, τη Γαλλία, το τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικό. Και υπάρχουν όμως άλλα μοντέλα στην Ισπανία, στη Γερμανία. Και δεν ε, υπολογίζουμε τον ίδιο τρόπο το ρίσκο. Υπολογίζουν τις πιθανότητες πιστοτικού ε, γεγονότος, χρεοκοπίας και στις περιπτώσεις του, των κρατικών ομολόγων. Και υπάρχουν επίσης διαφορετικές κατηγορίες ρίσκου ή buffer για τις ελληνικές τράπεζες που αναφερθήκατε πιο πριν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα ε, διακριτικής μεταχείρισης γιατί κάθε τράπεζα έχει το δικό της προφίλ ρίσκου. Κάθε χαρτοφυλάκιο, κάθε ισολογισμός πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Αυτό χρειάζεται προκειμένου να είμαστε και σκληροί και αυστηροί και ε, διαφανείς. Γιατί θέλουμε οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες να επιστρέψουν στις αγορές, ομολόγων και άλλε για να μπορέσουν να επαναχρηματοδοτήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ωραία και πάρει από το ΕΛΚ η Άστριτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Νουή. Εγώ λέω να μιλήσω γαλλικά την δική σας μετρική γλώσσα παρόλο που δεν είναι δική μου μετρική γλώσσα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι γαλλικά δεν θα εξασφανιστούν από τις συζητήσει περί οικονομικών, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θα αντικατασταθούν τα πάντα από τα αγγλικά. Χαίρομαι που επιλεγήκατε εσείς από άλλους υποψηφίου από τις διάφορες ευρωπαϊκές ε, αρχές και τράπεζες. Έχετε τα προσόντα. Είστε γυναίκα επίσης, που είναι, φαίνεται πιο σημαντικό για κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής, όχι τόσο για μένα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο ούτε το φύλλο, ούτε ο σεξουαλικός προσανατολισμός των διαφόρων υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν πιστεύω ότι σας επιλέξαμε επειδή είστε γυναίκα, αλλά εξαιτία των προσόντων σας. Τούτου λεχθέντος, εάν καλά κατάλαβα τις απαντήσεις σας, μου δημιουργήθηκε το εξή ερώτημα. Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της EBA μετά τη δημιουργία του SSM. Αν κατά δεν θεωρείτε ότι είναι περιττή πλέον η EBA. Αντιθέτως, λέτε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της. Ή μήπως θα έπρεπε να επαναξιολογήσουμε την εντολή της και τις αρμοδιότητες της, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη. Κοιτάξτε, ήρθα με το βιογραφικό μου ε, και όχι με το φίλο μου, τέλος πάντων, εδώ. Όσον αφορά το ρόλο της CBA, πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ουσιαστικός και Πιστεύω επίσης ότι θα προσανατολιστεί περισσότερο στα θέματα ρύθμισης, τεχνικά πρότυπα, ε, ε, συστάσεις, ε, κατευθυντήριες γραμμές για, τα, διάφορα θέματα τραπεζικά τέλος πάντων, για τα οποία ήδη έχει κάνει σημαντική δουλειά η EBA θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την EBA, το ενιαίο σύστημα, ο ενιαίος μηχανισμός. Η EBA θα συνεισφέρει στα stress test μετά την αξιολόγηση των ισολογισμών, αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα θετικό, στην ε, ομάδα υψηλού επίπεδου που έχει δημιουργήσει η ΕΚΤ e για την δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν ε, και εκπρόσωποι από χώρες εκτός ε, ενιαίου μηχανισμού σε διάφορα θέματα, ας πούμε για τις κοινέ ε, ομάδες εποπτείας ή στην αξιολόγηση των ισολογισμών. Θα πρέπει η στην αξιολογηση των ισολογισμων θα πρεπει η και η Ρία, να, ο Ανδρέα Ιρία να συμμετέχει ο υπεύθυνο δηλαδή τη CBA να συμμετέχει στις εργασίες μας, ε, γιατί πιστεύω ότι και η EBA και, το, και ο ενιαίος μηχανισμός, το SSM, πρέπει να ε, είναι παρόντα σε διεθνές επίπεδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε επίπεδο ενιαίας αγορές. Το, η αξιολόγηση των, των ισολογισμών θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ε, ευρωπαϊκές τράπεζες και η, η, η, αξιολόγηση θα γίνει των τραπεζών αυτών με βάση τα όσα έχει απαιτήσει η EBA. Η EBA ζητάει από τους, υπο, από τους επόπτες να κάνουν ε, ούτως ή άλλως μια αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών τους. Και οι μεγάλες ε, τράπεζες στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Γαλλία ε, ελέγχουν αν θέλετε και τις ε, εγχώριες τραπεζές τους. Ε, ε, στην Ανατολική Ευρώπη έχω έρθει σε επαφή με Πολωνούς συναδέλφους που μας είπαν ότι έχουν δύο τρόπους να δουλέψουν. Ή ασχολούμεθα με τις θηγατρικές των τραπεζών του ενιαίου μηχανισμού και κάνουμε μια ενιαία αξιολόγηση των, των ισολογισμών ή εμείς κάνουμε τη δική μας αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο και εσείς έρχεστε μετά και, το, και το, την επαναλαμβάνετε όσον αφορά τις θηγατρικές μέσα στα πλαίσια του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας. Είναι καλύτερο να τα κάνουμε μαζί τα πράγματα πιστεύω και αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, που βλέπουμε βλέπετε πώς ε, λειτουργούν καθημερινά οι επόπτες και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στην ενιαία αγορά, στην, στο single market δηλαδή, ε, στην EBA και στο SSM. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή το single market θα πρέπει να χάσει την σημασία του τώρα που μπαίνει σε λειτουργία το SSM. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές, κύριο Πιτέλα. Α, ευχαριστώ. Μία προειδοποίηση, αν θέλετε. Κυρία Νουή. Σχετικά με την έκθεση στο δημόσιο χρέος στα κρατικά ομόλογα. Να σας πω, από το 2007 Μέσω της αγοράς κρατικών ομολόγων οι τράπεζες έχουν παίξει έναν ρόλο συστηματικού σταθεροποιητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει μια σταθεροποίηση στην οικονομία. Τα κρατικά ομόλογα ήδη ε, είναι ένα κονδύλιο, του προπολογισμού ε, που μας επιτρέπει να ε, ελέγχουμε την κατάσταση της οικονομίας. Τα παράγωγα όμως βέβαια τώρα που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κάποιες τράπεζες στο Βέλγιο, στη Γαλλία κτλ δεν ε, εμφανίζονται με ιδιαίτερα σαφή και διάφανο τρόπο. Επί, επομένως, δεν πρέπει να χάσουμε τον στόχο μας. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τις, ε, τους, τις συναφείς κινδύνους. Η ερώτηση του κυρίου Μπάλσεν που έκανε πριν από λίγο, ε, να σας να τη συνεχίσω κι εγώ. Πόσο βλέπετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έκθεση στα παράγωγα, που αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα των τραπεζών. Δεν είπα ότι η έκθεση στα κρατικά ομόλογα είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλετε, στοιχείο του ενεργητικού των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Απλώς είπα ότι μέσα από την κρίση πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει, είδαμε ότι δεν υπάρχει ε, ακίνδυνο τελείως ε, στοιχείο του ενεργητικού. Και ε, ξέρουμε βέβαια ότι στο παρελθόν λέγαμε ότι σε μια υγιή οικονομία η αγορά κρατικών ομολόγων ήταν κάτι το οποίο δεν, ενέχει, δεν είχε κινδύνους. Τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα τοξικά προϊόντα στην αγορά ε, που κόστησαν πολλά χρήματα στις τράπεζες ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επόδυνη, επόδυνα ήταν θα έλεγα ε, όμως αντιμετωπίστηκαν αυτά, υπήρξαν κάποιες ε, ε, προβλέψεις, κάποιες, κάποιες ρυθμίσεις για αυτά τα legacy assets που είναι τα τοξικά προϊόντα τα οποία κληρονομήσαμε από την κρίση και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θα ε, αντιμετωπίσουμε. Στα στοιχεία αυτά θα ε, εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτή την αξιολόγηση του ισολογισμού. Ε, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, σε διάφοροι κανονισμοί που υιοθετήθηκαν σε, στις διάφορες χώρες, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά θα τα δούμε και κατά την άποψή μου έστω και αν υπάρχουν σαφείς διατάξεις ε, που μπορούν να πουληθούν τέλος πάντων ενδεχόμενα χωρίς ε, απώλειες. Ε, είναι η δουλειά του επόπτη να πείσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα προϊόντα αυτά. Διότι θέλουμε χώρο, αν θέλετε, στο, στον στους ισολογισμούς για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την πραγματική οικονομία. Και θα πρέπει ακριβώς όλα αυτά τα προϊόντα να φύγουν πρώτα. Ωραία. Εντάξει, σας ικανοποιεί η απάντηση. Άλντε. Ο Ραμόν Τρεμόσα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Μία ερώτηση για το δημόσιο χρέος. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα το πρωί Διάβασα το ίδιο άρθρο που ανέφερε και ο Αντολίν για τις επιπτώσεις ε, ε, της εποπτείας. Στη σελίδα 6 είναι δικό σας άρθρο. Όσον αφορά τα υψηλού επίπεδου ε, στοιχεία ε, ρευστότητας ε, θα, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να εκτεθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό συμβαίνει σε, πολλές ε, σε πολλά κράτη-μέλη. Στην Ισπανία που προέρχομαι για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ισπανικές τράπεζες έχουν μάνο από 300 δισεκατομμύρια ισπανικού δημοσίου χρέους, και αυτό αυξάνεται μήνα το μήνα. Δημιουργεί ένα τεράστιο αποτέλεσμα, δεν επιτρέπει να μπει τίποτα άλλο στους ισολογισμούς των τραπεζών. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δανειοδοτούν οι τράπεζες στην ουσία το δημόσιο τομέα κατά 10-15% και στο ίδιο ποσοστό μειώνουν την δανειοδότησή τους προς τον ιδιωτικό τομέα. Ερωτήσεις. Εάν λέτε ότι δεν έχει κίνδυνο το δημόσιο χρέο. Όπως λέτε, αυξάνει τα κίνητρα των τραπεζών να το κρατήσουν το δημόσιο χρέος. Άρα δεν δημιουργούμε πρόβλημα. Ότι έτσι δεν μπορούν να δανείσουν οι τράπεζες. Και στην επόμενη ανασκόπηση της ποιότητας του ενεργητικού όλες οι τράπεζες θα έχουν το ίδιο αρχικό επίπεδο ε, ε, αξιολόγησης. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει ότι και χώρες που έχουν τριπλό α και χώρες που δεν έχουν θα αντιμετωπίζουν, θα αντιμετωπίσουν τον ίδιο τρόπο. Εφόσον θέλετε να είστε η σιδηρά κυρία της εποπτείας θα πρέπει να πείτε κάτι συγκεκριμένο για να μας εξηγήσετε, να εξηγήσετε στους πολίτες μας και στους ψηφοφόρους μας περί πρόκειται. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τις ε, ανεπιθύμητες συνέπειες ενός πολύ στενού ορισμού των αρκετά ρευστών υψηλού επίπεδου στοιχείων του ενεργητικού και ε, ο διοικητή της Τράπεζα Γαλλίας και εγώ στη Γαλλία και οι συναδελφοί μου το έχουμε τονίσει επανειλημμένα. Νομίζω ότι χρειάστηκε χρόνος για να εισακουστούν οι απόψει μας διότι στην πρώτη εκδοχή του, στον πρώτο καθορισμό της αναλογίας ρευστότητας και ενεργητικού μάλλον ε, ρευστότητας και κάλυψης. Δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, τώρα έχουμε μια καλύτερη αναλογία. Είναι επαρκής αυτή η αναλογία. Για να μην αποτελεί υπερβολικό κίνητρο προς την έκθεση στο δημόσιο χρέος. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Αλλά αυτό καταφέραμε να επιτύχουμε μέσω των διαπραγματεύσεων. Δεν τα αποφασίζαμε μόνοι μας όπως φαντάζεστε θα εξακολουθούμε να ασχολούμεθα με το θέμα αυτό. Οι συζητήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για αυτήν την αναλογία ρευστότητας κάλυψης συνεχίζονται και επαναλαμβάνουμε επανειλημμένα την άποψή μας για να δούμε κατά πόσο θα βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά ήδη έχει σοβαρά βελτιωθεί. Μηδενικού κινδύνου τώρα αν υπάρχουν ε, τέτοια ρευστά στοιχεία ενεργητικού. Μόνο στην ε, τυποποιημένη προσέγγιση μπορεί να θεωρήσουμε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Μόνο στις μεγαλύτερες τράπεζες που είναι 85% των ε, τραπεζικών ενεργητικών του τομέα ισχύει κάτι τέτοιο. Και αυτές οι τράπεζες σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν δικά τους εσωτερικά μοντέλα για να υπολογίσουν αυτά, αυτούς τους λόγους και δεν έχουν έγκριση για να θεωρούν ότι είναι μηδενικού ρίσκου ε, τα κρατικά ομόλογα, μπορούμε να τους ζητήσουμε να αποτιμούν διαφορετικά από ό,τι θα ήθελαν ήδη να αποτιμήσουν αυτή την έκθεση. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πρώτου τεστ αντοχής, test που έκανε η EBA, υπήρξε στάθμιση του κινδύνου δεν ήταν ε, μηδέν αυτή η στάθμιση, αλλά ήταν ένα ελάχιστο όριο για τον υπολογισμό. Αυτά που τους έδωσε η EBA δεν έχουν αποφασιστεί όλα αυτά ακόμη, αλλά γιατί όχι, θα μπορούσαμε να έχουμε ελάχιστα επίπεδα για το ποια θα θεωρούμε ότι είναι τα σταθμισμένου κινδύνου στοιχεία του ενεργητικού, για να υπάρχει μια συνέπεια σε όλο τον τομέα. Γιατί αλλιώ πώς να εξηγήσει γιατί κάποιες τράπεζες μπορεί να θεωρούν ότι πρέπει να θέσουν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ για, ε, με τα οποία να μπορούν να καλύπτουν κρατικά ομόλογα και άλλοι 7 ή άλλοι 1,5. Γιατί ε, θα πρέπει να έχουν την ίδια αποτίμηση σε όλους τους ολογισμούς τα κρατικά ομόλογα. Αλλά δεν είναι μηδέν πρέπει βεβαίως να είναι στο σωστό επίπεδο. Αλλιώς ζητάμε κάποια buffer, δηλαδή κάποια μαξιλαράκια ασφάλειας για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επαρκές κεφάλαιο σε σχέση και με το προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας. Πρόεδρος, αν κατάλαβα, θεωρείται είτε ότι είναι σωστά αξιολογημένος ο κίνδυνος ή ζητάτε buffer για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν μόνιμες μερικές εξαιρέσεις για κάποιες μεγάλες τράπεζες. Νομίζω ήταν το άρθρο 145. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά κάπου εκεί δεν έχει πάει τώρα. Νουή, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ως ε, επόπτες, όπως οι συνάδελφοι στις διάφορες χώρες, εξετάζουμε το μοντέλο λειτουργίας της τράπεζας, να δούμε κατά πόσο ε, είναι στέρεο, ρωμαλαίο. Μετά βλέπουμε τι ποσοστό ε, κεφαλαιακών απαιτήσεων ζητάνε για τις διάφορες κατηγορίες συνεργητικού και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το ποσοστό κάλυψης, τότε ζητάμε επιπλέον buffer για να βεβαιωθούμε ότι έχουν επαρκές κεφάλαιο. Αυτό κάνουμε για το δημόσιο χρέος, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη έκθεση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών που είχαμε ορίσει στην αρχή. Τώρα υπάρχει ενδεχόμενο χρόνος, εάν κάποιος ε, θα ήθελε να θέσει κάποια ερώτηση. Κύριε Ανουή, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο. Θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση από αυτή που σας έκανα την προηγούμενη φορά. Έχετε μια ανδιαβισβήτητη εμπειρία στον τομέα που μας απασχολεί και προφανώς έχετε τα απαραίτητα προσόντα για να κάνετε τη δουλειά. Αλλά μια και είσαστε επόπτρια εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρέπει να είσαστε και στη Γαλλία όταν έλαβαν χώρα κάποια γεγονότα και ιδίως κάποια ε, τα οποία έθιξαν ένα τραπεζικό οργανισμό, χρηματοπιστωτικό οργανισμό που ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Βέλγιο, την Δέξια. Ε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιον ρόλο πιστεύετε ότι έπαιξε, είτε θετικό ή αρνητικό, η, αρχή, η η οργανισμο σας και Τι λάθο πιστεύετε ότι έγινε, γιατί όλοι είμαστε δικαιολογημένοι να κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Κοιτάξτε, τίποτα δεν έγινε. μέσω της εγκατάστασης της ING στην Γαλλία. Αυτό ήταν ένα λάθος που έκαναν κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί κάποιοι κάποια στελέχη της τράπεζας στο Λονδίνο ήταν ε, ε, ήταν στο ίδιο κτίριο με ε, κάποιο βρετανικό ίδρυμα το οποίο αντιμετώπισε προβλήματα. Δεν είχε καμία ανάμειξη η ING. Δεν θέλω να πω ποιος ήταν ο τραπεζικός οργανισμός που είχε πρόβλημα. Λοιπόν, συζητήσαμε την έκθεση στο, δημόσιο χρέος, στα κρατικά ομόλογα και πιστεύουμε και πιστεύαμε ότι υπήρχαν ε, κάποιες ε, ε, εκθέσεις στο δημόσιο χρέος και στα κρατικά ομόλογα τα οποία δεν παρουσίαζαν κανένα κίνδυνο. Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με την εταιρική διακυβέρνηση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι τράπεζες υπέφεραν λόγω της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης δεν εντοπίζονται. Τα εντοπίζουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά πολύ συχνά δεν έχουμε τους κατάλληλους κανονισμούς για να εφαρμόσουμε μία σωστή εταιρική διακυβέρνηση. Ελπίζουμε ευτυχώς ότι θα έχουμε αυτά τα εργαλεία σύντομα και για την φερεγγιότητα επίσης. Θα τα έχουμε τα εργαλεία αυτά και για το 34 και για το, τα εργαλεία φερεγγιότητας, ε, που είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά εργαλεία. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι όταν έχεις ομάδες κάπως περίπλοκες, ε, που είναι κατεστημένες σε διάφορες χώρες, ε, στην Ευρώπη ή όχι ή αλλού, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα διάφορα μοντέλα τα ε, εποπτείας τα οποία υπάρχουν και το μοντέλο της φιλοξενούσας χώρας είναι κάτι ε, το οποίο προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αλλά και αυτό δεν ήταν επαρκές για να ε, διασφαλιστούμε από προβλήματα που παρουσίαζει η οργάνωση και η λειτουργία μεγάλων ε, οργανισμών με διεθνή παρουσία. Αν σας καταλαβαίνω καλά, νομίζω ότι μου απαντούσατε στα γαλλικά, εκτός και τα γαλλικά των Βέλγων δεν σας ε, ικανοποιούν. Αλλά αν κατάλαβα καλά, η δέξια για την τέξια με τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας δεν έγινε κανένα λάθος. Άρα δεν, δεν, έχουμε, να μάθουμε δεν έχουμε να μάθουμε κάτι από το, από το πάθημά μας αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα απλώς ότι όπως και, και άλλοι και άλλοι επόπτες το γεγονός ότι η κατοχή δημοσίου χρέους, οι κρατικών ομολόγων ε, που από τις δημόσιες αρχές μπορεί να είναι, παρουσιάσει κάποιο κίνδυνο. Ε, αυτό τον κίνδυνο δεν τον αντιμετωπίσαμε επαρκώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αυτό είναι ένα λάθος ενδεχόμενα. Για το κόστος πιστεύω ότι οι Βέλγοι συνάδελφοι και εγώ εντοπίσαμε απόλυτα τα προβλήματα ε, ε, διακυβέρνησης, αλλά δεν μπορέσαμε να ε, επιβάλλουμε τις απόψεις μας, ίσως γιατί δεν υπήρχαν κανόνες γραπτοί, δεν υπήρχε κάποιο κείμενο, ίσως έπρεπε να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πυγμή. Αλλά τέλος πάντων, όπως σας είπα, ε, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια διμερή, τριμερή συνεργασία με τον ε, Λουξεμβούργο και ίσως αυτή η συνεργασία να μην ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Ίσως έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Τι να σας πω. Εδώ προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι η δεύτερη απάντηση ήταν καλύτερη από την πρώτη. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε εδώ η ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντανιέλ. Πρέπει να σε ευχαριστήσω επίσης γιατί μας έστειλες και τις γραπτές σου απαντήσεις εν γέρος. Έτσι όλοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν ε, την ε, ακρόαση. Πολύ καλή χειρονομία αυτή. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία. Αυτοί οι οποίοι δεν ε, ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποχωρήσουν. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα έχουμε μία σύντομη συζήτηση και θα βγει ένα ψήφισμα το οποίο θα περάσει στην Ολομέλεια που θα ψηφιστεί στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 5 Δεκεμβρίου και μετά θα περάσει από την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου με τη σύστασή μας. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί. Λίγα λεπτά μόνο διάλειμμα για να φύγει η Δανιέλ και οι άλλοι εξωτερικοί.